γη τους, γη εδώ και 300 χρόνια να ταξιδεύουν ελεύθερα στη χώρα τους και να εξαγάγουν τις ευρωπαϊκές ιδέες στην Ουκρανία. Ευχαριστώ κύριε Στογιάννοφ. Ο επόμενος, επόμενη μάλλον.